όπως ορίζονται αυτοί στα διάφορα ψηφίσματα. Έληξε η περίοδος συνόδου αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσοι δεν έρθετε στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, καλές